Okay. Point four of the agenda. Σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Έλεγχος στο κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων. Και σήμερα έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σχετικό ζήτημα για τα MRL, τις ελάχιστες απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων κτλ. Έχει ολοκληρωθεί, μάλλον ε, τρέχει η προπαρασκευαστική εργασία και θέλουμε να ενημερωνόμαστε πλήρως από την Επιτροπή και τα άλλα σχετικά σώματα, τα άλλα αρμόδια σώματα, γιατί εμείς ε, ελπίζουμε ε, σε μια καλή και ε, συνεπή ολοκλήρωση των εργαλείων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Να καλωσορίσουμε τον Patrick Πέρσον από την DG FISMA, τον Mark Adams από την ε, EBA. από την Τραπεζική Αρχή Θα αρχίσουμε με την Επιτροπή BA finally. και μετά την EBA και μετά... Κύριε Πίρσον, καταρχάς. Έχετε πέντε λεπτά έκαστος. Thank you, uh, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημαντικό σημείο έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Θα πω δύο πράγματα για το ΕΜΡΕΛ και μετά για το ΤΙΛΑΚ. Για το ΕΜΡΕΛ όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, η Κομισιόν ήδη ε, ενέκρινε το στάνταρ στις 23 Μαΐου. Εγκρίναμε τα προδιαγραφές που τροποποιούν την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ε, σε διάφορους τομείς. Με χαρά βλέπουμε ότι η Τραπεζική Αρχή συμφωνεί και δέχεται διάφορες τροπολογίες και πολλές μάλλον σε σχέση με αυτές που προτείναμε. Ένας τομέας όπου δεν ακολουθήσαμε την πρόταση, τις προτάσεις της τραπεζικής αρχής και αυτό ε, είναι εκεί που προτείνει να βάλουμε ένα μια εναρμονισμένη προδιαγραφή 8% για το MREL για τις συστημικά ε, συστημικές ε, τράπεζες τέτοιου τύπου. Για δύο λόγους δεν το κάναμε αυτό. Καταρχάς νομικός λόγος, η οδηγία είναι σαφής όσον αφορά την στάθμιση του MRL ότι δηλαδή πρόκειται για ειδική απέτηση ε, της τράπεζας ε, που ορίζεται ανά περίπτωση από τις αρχές εξιγίανσης Η εναρμόνιση ενός μήνυμου 8% δεν είναι θέμα του αν είναι αυτό επιθυμητό ή ανεπιθύμητο στο επίπεδο 2, είναι απλά παράνομο κατά τη γνώμη της Επιτροπής. Δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν εισήγαμε εναρμονισμένο μίνιμουμ 8% στι τεχνικέ μας προδιαγραφές είναι πολιτικής φύσης. Ε, και αυτό ανεφέρθη στου τριμερεί διαλόγους κύριε Πρόεδρε και συμφωνήθηκε ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή, να μην εναρμονιστεί ε, το συγκεκριμένο ε, θέμα στο επίπεδο 2. Οπότε αυτό αντικατοπτρίζεται σε αυτή την προδιαγραφή που σας προτείνουμε. Θέλω να είμαι σαφής. Συμφωνούμε ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα δυνατό MRL και το καταστέφουμε αυτό σαφές και προς, στην επιστολή μας προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ότι όλοι οι θεσμοί, όλες οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν ισχυρό MRL ώστε να μπορούν να είναι, να είναι δυνατόν να εξηγιανθούν. Δεν υπάρχει διαφωνία εδώ, απλώς δεν υπάρχει δυνατότητα να αναρμονιστεί αυτό σε πράξη επίπεδου 2. Τώρα, αυτό τι αλλάζει στο κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ε, όχι, δεν αλλάζει τίποτα στην πράξη, διότι οι αρχές εξυγένσης ε, έχουν τη διακριτική ευχέρεια στο κείμενο επίπεδο 1 στην ε, σχετική οδηγία να θεσπίζουν το MREL στο κατάλληλο επίπεδο που μπορεί να είναι κάτω από το 8% αλλά μπορεί να είναι και πολύ ψηλότερο από το 8%. Αυτή η διακριτική ευχέρεια ε, αφήνεται στην αρχή εξυγίανσης ανά τράπεζα, ανά περίπτωση. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, Πρόεδρο, όσον αφορά το σχέδιο προδιαγραφών. Το Κοινοβούλιο έχει τρει μήνε για να φέρει τι αντιρρήσει του. Ξέρουμε ότι οι αρχέ εξηγήσει θέλουν γρήγορα να προχωρήσουν και να ορίσουν του ε, στόχου MRL γρήγορα και ελπίζουμε το, το Κοινοβούλιο επίση να συμφωνήσει να μην καθυστερήσει την έναρξη ισχύω αυτών των τεχνικών κανόνων. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, γιατί δεν είναι εδώ το τέρμα. Όπως γνωρίζετε η Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα συντάξουμε νομική πρόταση ε, για να εισαχθεί το TILAC στην κινητική νομοθεσία. Αυτό τροποποιεί την ισχύουσα νομοθεσία επίπεδου 1. Θα έχουμε πλήρη πρόταση της Επιτροπής και το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο θα έχουν πλήρη νομοθετική αρμοδιότητα να βελτιώσουν, τροποποιήσουν, σχολιάσουν ε, την εν λόγω πρόταση. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να υποβάλουμε την πρόταση μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο μέχρι σήμερα σε τεχνικό επίπεδο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και ε, μέσα σε αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να βρούμε μια λογική και αποδεκτή λύση ανάμεσα στο τι έχει συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για το ΤΙΛΑΚ και για το πώς θα μπορούσαμε αυτό να το εφαρμόσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ε, τροποποιητικής νομοθετικής πρότασης. Όπως σας είπα, σκοπεύουμε να υποβάλουμε μέχρι το τέλη του έτους νομοθετική πρόταση. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε ρυθμιστικές απλοποιήσεις. Δεν πιστεύουμε ότι οι τράπεζες μας θα πρέπει να υπόκειται σε δύο διαφορετικά στάνταρ, τα έμερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και τα TILAC στο παγκόσμιο επίπεδο ταυτόχρονα. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μέχρι τα τέλη του χρόνου και να την περιλάβουμε στην πρότασή μα. Τα MRL και τα TILAC έχουν την ίδια, ε, τους ίδιους στόχους. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις προδιαγραφέ τη διεθνής με τις ευρωπαϊκές και θα σταματήσω σε αυτά γιατί μου δώσατε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω κάποιες ε, ερωτήσεις για σας, αλλά θα τις κάνουμε αργότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τώρα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ σήμερα μετά από την έγκριση από την Κομισιόν των Εμιρέλ αλλά και των άλλων τεχνικών προδιαγραφών που έχουμε ε, προετοιμάσει στο πλαίσιο του BOD και πολλά από αυτά τα καταθέσαμε τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Τώρα προχωράει η διαδικασία επικύρωσης. Ε, πιστεύουμε ότι είναι άλλο ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του νέου καθεστώτος των τραπεζών, εξυγίανσης των τραπεζών. Τα MRL είναι πολύ σημαντικά, σημαίνει ότι οι αρχές εκαθάρισης ε, μπορούν να αρχίσουν να ε, ολοποιούν, να ολοκληρώνουν τις μεθόδους τους για τα MRL και κατόπιν να λάβουν τις επιφάσεις, αποφάσεις ε, μέχρι το τέλος του έτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια η ολοκλήρωση αυτών των πολιτικών περιμένει ε, την επικύρωση των προδιαγραφών. Αυτό είναι ένα εμπόδιο για να προχωρήσουμε. Συμφωνήσαμε με την ε, Κομισιόν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε το σύντομο των δυνατών και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να προσφέρουμε όποια βοήθεια θέλετε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ελέγχου και τον Εμιρέλ. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες που ενέκρινε η Κομισιόν στις δικές μας τις προδιαγραφές, συμφωνούμε με την Κομισιόν ότι αυτά δεν θα οδηγήσουν σε σημαντικές πρακτικές αλλαγές στη διαδικασία αξιολόγησης των Εμιρέλ. Κατά την άποψή μας ε, δεν υπάρχουν εκατότατα όρια, ούτε πρέπει να υπάρχουν. Ε, πιστεύουμε ότι το bail είναι 8% πριν φτάσει κανείς στο Ταμείο Εξυγείωνσης και στην περίπτωση που δεν αρκούν οι διπόλοι της τράπεζας, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στον ορισμό των Εμιρέλ. Να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στους ενωσιακούς κανόνες ε, για το τι μπορεί να συμβεί τώρα και πώς οι αρχές εξυγίανσης θα το ανακοινώσουν αυτό στις τράπεζες. Βλέπουμε ότι πολλές αρχές εξυγίανσης συμφωνούν με αυτό, άρα δηλαδή η πρακτική διαδικασία μπορεί να προχωρήσει ε, όπως είχε σχεδιαστεί. Εξάλλου, συμφωνούμε απόλυτα με τη δουλειά της Κομισιόν έτσι ώστε να υπάρχει μια νομοθετική πρόταση ε, για τα SPD standards και εμείς ε, όταν συντάσσουμε τα κριτήρια για τα MRL κατ' ουσίαν έχουμε κατά νου ε, το μέλλον όπως το είχε προγραμματίσει η FSB και θεωρούμε ότι οι μεγάλες τράπεζες ε, θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για το ΤΙΛΑΚ όπως και για το εμιρέλ, Γιατί είναι σημαντικό οι τράπεζες να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές για τον ίδιο στόχο. Όπως ε, ήταν ήδη σαφές, ε, η σημαντική διαφορά ανάμεσα στα ΤΙΛΑΚ και τα MRL είναι ότι τα Μιρέλ αφορούν περίπου 7.000 πιστοτικά ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ε, πιο ε, σημαντικό γιατί το TILAC αφορά λιγότερους. Άρα δηλαδή στο πρώτο πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Όσον αφορά την εφαρμογή των TILAC, ε, κάποια στοιχεία του TILAC θα πρέπει να ισχύουν και για τα Μιρέλ. Ακούμε από τις αρχές καθάρισης ότι η τατίλακ, ε, δημιουργούν κάποια πρακτικής φύσεως θέματα. Είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να προχωρήσει γρήγορα με ε, σαφή καθοδήγηση στις τράπεζες για το τι πρέπει να περιμένουν ως τελικές απαιτήσει για τα TLAC ή τα MIREL, έτσι ώστε οι τράπεζες να αρχίσουν να ε, προγραμματίζουν, να κάνουν τα προγράμματά τους ε, για τα επόμενα 3-5 χρόνια κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Επίσης, ε, κάτι άλλο που μας ανησυχεί από κάποιες άλλες αρχές έχει σχέση με το πώς τα MRL θα εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι τράπεζες ε, να μπορούν να καθαριστούν και ε, βεβαίως θα δούμε τις προτάσεις Κομισιόν έτσι ώστε να διαπιστώσουμε ότι όλα αυτά είναι και συμβατά με τη δική μας την εντολή. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να συμβάλλουμε στην ε, συζήτηση για την εφαρμογή των ΤΙΛΑΚ είναι αρχές καλοκαιριού να υποβάλουμε μια ενδιάμεση έκθεση ε, επειδή η εφαρμογή των Emerald είναι πολύ αρχική για θέματα όπως είναι κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσει, εμείς δεν θα μπορέσουμε ε, να τα εξετάσουμε όλα, αλλά έχουμε ε, καλύψει, έχουμε συγκεντρώσει δεδομένα από 120 τράπεζες και επίσης έχουμε εξετάσει και τις ε, πολιτικές ε, που έχουν καταθέσει οι αρχές ε, καθάρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλες αρχές που ασχολούνται με το ΤΙΛΑΚ στην Ελβετία, στις ΗΠΑ και αλλού. Και με βάση αυτά θα έχουμε ενδιάμεση έκθεση για τεχνικά θέματα. Θα δούμε και θέματα κοινοποίησης στοιχείων ε, γιατί εκεί προκύπτουν τέτοια θέματα όπως ε, και στον πυλώνα 2 ε, σας είπα ότι θα πρέπει να κοινοποιούνται στοιχεία που είναι σημαντικά για τους επενδυτές και σε επίπεδο MRL και σε πολιτικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, καταρχάς ε, να πω το προφανές. Είναι πολύ σημαντικός ο καθορισμός του NMRL για να είναι φερέγγιες οι τράπεζες. Και είναι σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για να συζητήσουμε σήμερα αυτό το θέμα. Θα πρέπει να δούμε ίσως γιατί είναι τόσο σημαντικό να έχουμε αυτές τις ελάχιστες απαιτήσει ε, για να μπορέσει το bail-in να είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο εξυγίανσης, όχι bail-out δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν αποδεκτές υποχρεώσεις. Και όταν μια αρχή εξυγίανσης θεωρεί ότι πληρούνται προϋποθέσεις εξυγίανσης, θα μπορεί μετά να μετατρέψει το χρέος και τα λοιπά ή να κάνει κάτι άλλο. Αυτό ήταν ο ορισμός και το είπαν και οι προλαλήσαντες ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε σε ένα συστημικό αποτύπωμα του ε, φορέα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι γενικό που να ισχύει για όλους. Ε. Ένα MRL 8% αλλά αυτό θα είναι το κατώτατο, για πολλές θα είναι μεγαλύτερο για τις μεγαλύτερες τράπεζες της Τραπεζικής Ένωσης, αναφέρουν. Και εγώ μιλώ για τις τράπεζες που είναι υπό την εντολή του SRB. Κυρίως. Δεν εστιάζω δηλαδή σε όλες τις τράπεζες της Τραπεζικής Ένωσης. Για αυτές λοιπόν που είναι στη δική μας εντολή, Νομίζω ότι είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι αν υπάρξει πρόβλημα, η εξηγένση θα είναι η καταλληλότερη λύση, 8% δηλαδή. Ε, λογικό. Τώρα, ατομικός καθορισμός MRL, αναόμιλο ή ανατράπεζα, θα πρέπει να ακολουθείτε μια προκαθορισμένη διαδικασία, η ανατραπεζα θα πρεπει ξεκίνησε ήδη φέτος σε επίπεδο ε, ομίλων γελούσα πριν, διότι έχουμε τώρα τα πρότυπα, αλλά δεν σημαίνει ότι την άλλη Δευτέρα θα έχουμε λάβει όλες μας τις αποφάσεις. Είναι λίγο πιο μακρά αυτή η διαδικασία. Και αυτή τη στιγμή ε, το Συμβούλιο συλλέγει στοιχεία από την Κομισιόν, το SRB, για να προετοιμάσει αυτές τις ε, αποφάσεις, το ενίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Έχουμε συζητήσει επίσης ε, την κατευθυντική αυτή πράξη ε, και το Συμβούλιο εξηγήσει τα παρακολουθεί ε, τα πράγματα και δεν βλέπει αυτή τη στιγμή το παρόντος ανάγκη να αλλάξει πολιτική λόγω της έγκρισης αυτών των κανόνων. Είναι καλοδεχούμενη η σαφήνεια της έγκρισης αυτής της κατεξουσιοδότησης πράξης για τον καθορισμό των MREL, των βασικών ενιών, για τις αρχές ε, και για τον κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει πλέον αναφορά στον ελάχιστο στόχο το 8% γιατί σε συστημικά σημαντικές τράπεζες διαγράφει και αυτή η αναφορά όπως και το, λεγόμενο περίοδο, την τυποποιημένη περίοδο phase-in. Υπάρχουν και νομικοί λόγοι που δεν θα επηρεάσουν όμως τις αποφάσεις του Συμβουλίου Εξυγίανσης τώρα στο διεθνές πλαίσιο για να περάσω στην TILAC τη συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών. Αυτό είναι ένα πρότυπο που ανέπτυξε το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα FSB και έχει γίνει δεκτό και από το G20. Χρειάζεται μεγάλη δυνατότητα απορρόφηση βέβαια, τουλάχιστον του 16% ε, των περιουσιακών στοιχείων και 6% του συνολικού ποσοστού ε, μόκλευσης από το 2019 και θα ανεβούν τα ποσοστά αυτά μέχρι το 2022. Κάντε εσείς ε, αριθμητικές πράξεις να περάσετε τα μήνυματα, αλλά τέλος πάντων. Το TILAC e εφαρμόζεται άμεσα. Αυτό δεσμεύτηκαν να το πράξουν οι G20, όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις ε, για πρότυπα του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. λέει και έμερα είναι σημαντικά βήματα για τη δημιουργία ενός ότιμου πεδίου ανταγωνισμού για τις τράπεζες. Θα δοθούν σαφή κίνητρα για μεγαλύτερη φεργιότητα και δυνατότητα ε, εξυγίανσης. Και δεν θέλουν ποτέ να έχουμε τελικά μια τράπεζα too big to fail. Το bail-in και όχι το bail-out πλέον θα είναι ο κανόνας. και έχουμε και αυτό το 8% που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα ίδια κεφάλαια και τις αποδεκτές υποχρεώσεις πρώτα. Προσπαθώ να μην είμαι τόσο γρήγορη όταν ε, μιλάω, ε, ή μάλλον όταν διαβάζω, αλλά μάλλον ήμουν πιο γρήγορη την προηγούμενη φορά. Πώ θα εφαρμόζεται το MRL και TILAC. Θέλουμε να εφαρμόζονται συμβατά μεταξύ του, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ευρωζώνη, εντό Ευρωζώνη, μάλλον εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά θα πρέπει εμεί τώρα να εφαρμόσουμε το Συμβούλιο Εξήγηση αυτή, ε, τι ε, αρχέ αυτέ. Αυτή είναι η νομική απέτηση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση το ΤΙΛΑΚ. Δεν είναι κρίμα αυτό. Δεν βλέπω να υπάρχει, ελπίζω τουλάχιστον, σύγκρουση, αντιπαράθεση. Εμεί εργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με άλλου στην ομάδα εργασία Προς το παρόν όμως εγκρίνουμε τα Emerald και λαμβάνουμε αποφάσεις για τα Emerald και έπειτα θα συμπεριλάβουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της στήλα σε αυτές τις αποφάσεις. Για να αντιμετωπίσουμε και άλλα εμπόδια εξυγίανσης. Αυτός είναι ο στόχος μας ε, για το 16 και πιο Και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας ε, είπατε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Χόκμαρκ. Ευχαριστώ πολύ και όλα αυτά που ακούσαμε. Ευχαριστώ για αυτά. Ε, να το πω έτσι πολύ ήπια. Για μένα αυτά όλα είναι πολύ περίπλοκα. και βλέπω ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση, άλλη αυτή της Κομισιόν και άλλη της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Νομίζω όμως ότι θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις τελικά πώς ακριβώς επηρεάζουν το επίπεδο των Εμιρέλ, δηλαδή με ποιον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο MRL όταν αυτό είναι απαραίτητο για το Μπέιλιν. Και δεύτερον, αυτοί οι δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης ε, του προβλήματος πώς ε, ακριβώς ε, επηρεάζουν το τίλακ και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ε, προετοιμάσουμε ένα τίλακ που θα έχει πιο άμεση επιρροή στις ε, τράπεζες. Εξ όσων κατάλαβα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το 8% δεν το θεωρεί νόμιμο, αλλά είναι αυτή η άποψη και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Ε, και αυτή είναι μια ερώτηση. Βέβαια, την κατεξοδότηση πράξη πρέπει να συζητήσουμε λίγο παραπάνω, αλλά τουλάχιστον η απάντηση αυτών των ερωτήσεων θα μπορούσε εμένα να με βοηθήσει ε, στη συζήτηση. Η Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους ε, τρεις ε, θεσμούς που έλαβαν το λόγο, γιατί από ό,τι φαίνεται στο επίκεντρο ε, της διαδικασίας έχουμε σοφούς ανθρώπους και σοφούς θεσμούς. Και αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, διότι προχωράμε σε πολύ περίπλοκα πράγματα. Είναι η πρώτη φορά ε, που μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα ύδατα και χωρίς τη βοήθεια, μάλλον εγώ ε, θυμάμαι που προσπαθήσαμε με τον ε, εισηγητή και τους συνεισηγητές να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που δεν πρέπει, που δεν είναι να αποτύχει. Μπήκαμε, όπως σας είπα, σε χαρτογράφητα νερά και τώρα πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερε ικανότητες, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην προκύψουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Και αυτά έχουν κυρίως σχέση με το γεγονός ότι όταν υπολογίσαμε ένα 8%. Η βασική μας ανησυχία ήταν να εγγυηθούμε ότι στην επόμενη κρίση οι φορολογούμενοι δεν θα κληθούν να στηρίξουν ε, καταραίουσες τράπεζες. Αυτό βέβαια συζητήθηκε μεταξύ μας και καταλήξαμε στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα 8% bail-in σε όλους τους θεσμούς ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το επιχειρηματικό τους μοντέλο γιατί δεν είχαμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Ακόμα και με την κρίση δεν υπήρξε της τάξης του 8% ούτε στην Ευρώπη ούτε στις Ηνωμένε Πολιτείες. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα που περνάμε στη φάση της εφαρμογής οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάνουμε το σωστό και να μην καταλήξουμε σε ανεπιθύμητες συστημικές επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν είτε από έναν συστημικό οργανισμό που θα καταρρεύσει είτε από σε μη συστημικά παραδοσιακά στοιχεία που οι πολίτες γενικά τα θεωρούσαν ιδιαίτερα ασφαλή. Είναι λοιπόν ε, πολύ επικίνδυνο να έχουμε ανεξέλεγκτη κατάρρευση μεγάλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο αυτό από ένα παραδοσιακό ε, μοντέλο το οποίο λέει bail-in μεγάλων χρεών, δανείων. Το θέμα είναι ότι πρέπει ε, να επιστήσουμε την προσοχή σας σε αυτή τη διαδικασία και όλων των υπόλοιπων εταίρων να διευκρινίσουμε ότι ακριβώς χρειάζεται διευκρινίση για να μην ε, προκληθούν συστημικά προβλήματα και να μην τεθεί ε, σε κίνδυνο όλο αυτό το σχήμα που έχουμε ήδη διαμορφώσει. Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνοντας Εμιρέλ και Τιλάκ υπάρχουν διαφορές, μερικές είναι ε, σαφείς, αλλά εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι υπάρχει μια διαφορετική μεταβατική περίοδος και πάνω απ' όλα το τιλάκ. δεν ισχύει παντού σε αντίθεση με τα Μιρέλ και μιλάμε για περίπου 6.000 θεσμούς στην Ευρώπη. Στην ε, Τραπεζική Ένωση, καταλήγοντας, θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε ε, για να κατανοήσουμε τη λύπη στο μοντέλο αυτό και τέλος για να διευκρινίσουμε αυτό που λείπει έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο όλο αυτό που έχουμε κάνει απλά και μόνο γιατί δεν βρήκαμε τις λεπτομέρειες. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν που ανέλαβε την πρωτοβουλία και ελπίζω η Κομισιόν ε, να ε, προβάλλει τις αποφάσεις ε, πρώτου επίπεδου. να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες για να ορίσουμε τι είναι τα διαφορετικά εμιρέλ, να επεξεργαστούμε το μοντέλο ε, με την πάροδο του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ και λυπάμαι που ε, κατανάλωσα λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν βλέπω να υπάρχουν ε, σκιώδεις στον ECR. Για τους φιλελεύθερους παρακαλώ. Ευχαριστώ η κυρία Σελβί Γκουλάρη. Ήταν πολύ καλό που ακούσαμε την Κομισιόν. Ε, χαιρετίζω την κυρία Κένινγκ. ε, και επίσης όλους οι υπόλοιπους. Με τη δική μου έκθεση πριν από κάποιες εβδομάδες το Κοινοβούλιο επέβαλε μια έκθεση που θέτει το θέμα της σχέσης μας με τους παγκόσμιους διεθνείς οργανισμούς που ορίζουν κανόνες. Και αυτό που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε ήταν να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες ποιος αποφασίζει σας καλώ λοιπόν να διερωτηθείτε αν το Financial Stability Board έχει το τελευταίο λόγο, ας το κλείσουμε εδώ το μαγαζί γιατί υπάρχουν ε, υπουργοί, υπάρχουν ε, ε, κεντρικοί τραπαζίτες, αλλά κανένας εκπρόσωπος των πολιτών. Με όλο το σεβασμό δε που έχω και για το ΖΕ20 και το τι έκανε στη διάρκεια της κρίσης, ότι και εκεί υπάρχουν χώρες, περιλαμβάνονται χώρες που δεν είναι και πρότυπα δημοκρατίας και θα πρέπει ίσως να διερωτηθούμε, ε, γιατί εντάξει δεν μπορούμε να λέμε έρχεται από το J20, άρα είναι καλό. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε δηλαδή σαν να ήταν ε, Ευαγγέλιο τα όσα μας λέει το G20, όπως είπε και Ελίζα. πούμε για το πεδίο εφαρμογή ε, υιοθετούμε τη λογική των Αμερικανών που συχνά δεν παίρνουν μέτρα και παρά μόνο για ορισμένο ε, θεσμούς εδώ είτε για άλλα κείμενα, είτε απευθυνόμαστε στο σύνολο του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα που είναι τελείως διαφορετικό. Σε ορισμένε χώρες όπως η δική μου θέλω να σας τονίσω ότι δεν είναι οι μεγάλες τράπεζες που σήμαναν κίνδυνο για την κρίση. Αυτές ήταν πολύ καλά εποπτευόμενες και δεν ε, χρειάστηκε να γίνει bailout για αυτέ Ενώ σε άλλες χώρες είχαμε να κάνουμε, ε, να, να, να χρειάστηκε να ζητήσουμε από τον φορολογούμενο. Και έπειτα πρέπει να διαβάσουμε τα κείμενα. Η οδηγία λέει σαφώς ότι η προσφυγή στο MRL, στο κανόνα του 8%, πρέπει να ερμηνεύεται αναπερίπτωση. Και ότι για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στα κονδύλια, και όχι ότι εξορισμού είναι ο κανόνας, όταν λέει ότι πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια, increase clarity, αυτό δεν σημαίνει ότι εφόσον υπάρχουν περιθώρια εκτίμησης ότι τελικά εφαρμόζουμε τον ίδιο κανόνα για όλους, γιατί αυτό σημαίνει ότι υποκαθιστούμε τον νομοθέτη. Σίγουρα δεν είχατε σκεφτεί αυτό και ίσως θα μπορέσουμε εκεί να συμφωνήσουμε. Τελευταίο θέμα. Εγώ διαρωτάμε αν δεν υπάρχει ηθικός κίνδυνος σημαντικός. Γιατί να μπορούμε έτσι να έχουμε πρόσβαση στο Ταμείο Εξυγίασης. Δεν ήταν αυτό που είχαμε σκεφτεί και σκέφτομαι και τα σχόλια της Ελίζας ε, και των υπολείπων. Ότι δηλαδή θέλαμε να φτιάξουμε ένα κείμενο που να λέει ότι όχι από τη στιγμή που έχει κάνει δυσκολίες θα έχει πρόσβαση και στο ταμείο. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ πολύ σοβαροί σε αυτές τις πτυχές, να μην μπούμε σε χωράφια όπου δεν θέλει ο νομοθέτης να μπούμε και να θυμηθούμε και την ε, νομολογία Μερώνη που που λέει ότι όλες οι ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκοί οργανισμοί θα πρέπει να εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανόνες και όχι για να δημιουργούν νέους, γιατί αυτό μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία μας, γιατί γι' αυτό μιλάμε τελικά. Όλοι συμφωνούμε να πλαισιωθεί η δραστηριότητα η τραπεζική, δουλέψαμε όλοι σκληρά γι' αυτό, αλλά δεν θέλουμε τελικά και οι τράπεζες να μην μπορούν να δουλέψουν και να λειτουργήσουν. Ευχαριστώ. Merci, Yes, uh, good evening everyone. Uh, Λάμπερτς. Ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Ναι, και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε η Σιλβή, τους ρόλους του καθενός δηλαδή, όπως ε, η, η, και ότι οι νομοθέτες ε, πρέπει να αποφασίσουν και όχι αντιστρόφως ανάλογα. Σελβί μπορεί να μην χρησιμοποιήσετε πολλά χρήματα των Γάλλων φορολογούμενων, αλλά σίγουρα αν οι Αμερικανοί δεν είχαν σώσει την ε, AIG, τότε η Société Générale, μου φαίνεται, της Γαλλίας θα είχε και εκείνη ε, βουλιάξει. Είναι λεφτά φορολογούμενων και αυτά και α μην είναι το άλλο φορολογούμενων. Τώρα, άκουσα πολύ προσεκτικά την Κομισιόν και τα επιχειρήματά της. Εσείς αναφέρατε δύο επιχειρήματα, ε, το νομικό και το πολιτικό. Εγώ πιστεύω πως το νομικό επιχείρημα ήταν γραμμένο με ψηλά γράμματα, ενώ το πολιτικό με πολύ επιχείρους ε, χαρακτήρες, γιατί όλα αυτά είναι πολιτικής φύσης. Εγώ είμαι απλό άνθρωπος, δεν είμαι νομικός, αλλά ξέρω ότι εμείς οι νομοθέτες γράψαμε πως αν θέλει να έχεις πρόσβαση στο Ταμείο Εξυγένσης πρέπει να έχεις ενσωματώσει το 8% των συνολικών ζημιών και αυτό είναι γραμμένο στην νομοθεσία. Τώρα ειλικρινά μπορείτε να μου πείτε ότι οποιοδήποτε συστημικό ε, ε, ίδρυμα που θα πρέπει να εξηγενθεί δεν χρειάζεται να πάει στο Ταμείο Εξυγένσης δεν θα πάει απαραίτητο μάλλον από εκεί. Μα δεν μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο. Ξέρετε ότι εφόσον υπάρχει ένα συστημικό σεσμό που πρέπει να πάει να εξυγιανθεί, θα πάει στο Ταμείο Εξυγίανση. Οπότε βεβαίω και χρειάζεται ένα ποσοστό. Ένα έμρελ με συγκεκριμένο ποσοστό είναι προφανέ. Και δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι το νομικό σας επιχείρημα θα σταθεί. 30 δευτερόλεπτα στο 10 εάν χρειάζονταν να διαβάσει ολόκληρη την νομοθεσία και να πει ναι, χρειάζεσαι 8% μπέιλι να μαθες να έχεις πρόσβαση στο ταμείο. Οπότε η πρόθεση του νομοθέτη είναι ξεκάθαρη. Εγώ πιστεύω πως ε, εδώ παίζεται με ένα νομικό παιχνίδι μόνο και μόνο για να υπακούσετε στις πολιτικές πιέσεις. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία των όσων κάνετε. Ειλικρινά λοιπόν, εγώ είμαι με την ε, τραπεζική αρχή εδώ δεν νομίζω δεν θυμάμαι τώρα τη διατύπωση που χρησιμοποίησε η Σιλβία, ότι βασικά δηλαδή κάνουν, ε, ε, βασίζονται με την νομοθεσία για να προβούν σε φάνταστες λύσεις. Όχι, εγώ λέω πως εκεί διάβασαν πολύ καλά και μόνο ένα συμπέρασμα μπορεί κανείς να βγάλει. Και βέβαια μπορεί να πάει ανά, ανά, ανά περίπτωση, αλλά πάντα θα είναι πάνω από το 8%. Μπορεί να είναι δεν λέει ότι δεν μπορείς να πας ανά τράπεζα αν υπάρχει ένα όριο 8%. Και πάλι το νομικό σας επιχείρημα είναι σαθρό. Τώρα, για το τίλακ, τα καλά νέα είναι ότι αν επιβάλλουμε το 8% συνολικών ζημιών ως μίνιμουμ απέτηση για επιλεξιμότητα για τις συστημικές τράπεζες, ε, θα τηρούν και το τίλακ. Θα τηρείται και το τίλακ, θα ικανοποιηθεί και το τίλακ. Αν κάνουμε το ένα λοιπόν, καλύπτουμε και το άλλο, οπότε χτυπάμε ε, δύο στόχους με, με, μία, με τη μία. Και τώρα, όλα ωραία και καλά να λέμε ότι θέλουμε ότι θέλουμε να καλύψουμε τους φορολογούμενους, αλλά αυτοί που, θέλουν να που δεν θέλουν να πληρώσουν είναι οι, φορο... οι μέτοχοι. Λένε, κάνουν ένα σωρό νοησίες. Οι μέτοχοι καταλήγουν στο να πληρώνουν τη ζημιά και αυτό είναι καλό. Ναι, αυτό αποφασίσαμε, ότι το υπερβολικό το πλεόνασμα κεφαλαίου σε σχέση με τα νεζονικές υποχρεώσεις πάει προς το MRL. Και επιμένω να μην το αποδυναμώσουμε αυτό, Περιμένω, ε, επιμένω όπως εκείνοι που λένε ότι για να ξεφορτωθούμε όλες αυτές τις δυσκολίες θα πρέπει να έχουμε πολύ ψηλότερες κεφαλαϊκές απαιτήσει και να ε, βασιστούμε σε ποσοστά μόχλευσης και, και όχι σε αυτά εδώ τα τελείωσα ασταθήκια βέβαια. Ευχαριστώ. Σας ε, συστήνω να διαβάσετε το χειρόγραφο του Κωνστάντσιο ε, στο κοινοβούλιο που κατά την άποψή μου ε, θα σας δώσει μια σαφή εξήγηση γιατί το 42 και το 44 είναι τελείως διαφορετικά. Δεν βλέπω άλλες πολιτικές ομάδες. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Μπάλτς είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ τη συζήτηση ε, σήμερα τη βρίσκω πάρα πολύ σημαντική γιατί τα πλεονεκτήματα της Τραπεζικής Ένωσης είναι ακριβώς ε, στο μέλλον ο φορολογούμενος ε, να μην ευθύνεται σε περίπτωση κατάρρευσης της τράπεζας. Τώρα πρόκειται για τη δυνατότητα εξυγίανσης των τραπεζών και μετά από τα λόγια πρέπει να ακολουθήσουν πράξεις. Αν δούμε λοιπόν τις ε, νομικές υποχρώσεις και τις δικές μας, να υπάρχει ένα σταθερό καθεστώς Μπέιλιν, αυτό σημαίνει ότι το 8% στον πυλώνα 1, κατά την άποψή μου, είναι απολύτως απαραίτητο. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υλοποιεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Εξυγήνης, αυτό με ανησυχεί. Η εφαρμογή του ΤΙΛΑΚ πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό καθεστώς εξυγίανσης και γι' αυτό το λόγο εγώ σήμερα θα ήθελα να διατυπώσω κάποια ερωτήματα εφόσον πολλοί συνάδελφοι είπαν πάρα πολλά και έξυπνα. Ερωτώ την Κομισιόν. Η Κομισιόν προτίθεται να δώσει ουσιαστικές αρμοδιότητες ε, στην αρχή εξυγίανσης ε, και κυρίως να εφαρμόζεται μοιρέλη στον πυλώνα 2. Κατόπιν θα ήθελα να γνωρίζω ε, όσον αφορά την subordination η Κομισιόν και την, το, η Ευρωπαϊκή Αρχή τι ακριβώ πιστεύουν ότι τα μοιρέλη στον πυλώνα 2 θα πρέπει να ζητούν απαιτητικά την ε, subordination και πώς ακριβώς ε, πρόκειται να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Και τελευταίο ερώτημα, το TILAC επιτρέπει δυνατότητα εξαίρεσης 3,5% από το αίτημα τους, ε, της subordination. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται να συμπεριλάβει αυτό το δικαίωμα της αρχής της ε, στην ε, νομοθεσία και στις νομοθετικές διατάξεις που θα προτείνει. Υπερβάνς έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την σημερινή συζήτηση και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Εγώ έχω τρία βασικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι η Κομισιόν λέει ότι θα μας φέρει καινούριε προτάσεις για το ΤΙΛΑΚ. Και όσον αφορά τη συνοχή της εφαρμογής, ειλικρινά διερωτώμεθα. Γιατί να μην έχουμε βάλει τα δύο κείμενα παράλληλα, να δούμε ποιο είναι το καλύτερο είναι μια αγαθή ερώτηση, ε, σχεδόν ανόητη. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει στενή συσχέτιση μεταξύ των δύο. Εάν δεν κάνουμε λοιπόν τα δύο ταυτόχρονα, κινδυνεύουμε να είμαστε συνεπείς. Εκτός αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το T-Lag για να δούμε τις ασυνέπειες του MRL. Δεν νομίζω πως μπορεί ο Ευρωπαίος νομοθέτης να ακολουθεί μια τέτοια στρατηγική. Πώς θα εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι τα όσα συμφωνούμε εμείς σήμερα θα είναι όντως, θα ληφθούν μάλλον όντως υπόψη στη στιγμή της έναρξης ισχύω εντός της Ένωσης του ΤΙΛΑΚ, επί τη βάση της πρότασης της Κομισιόν. Το δεύτερο είναι ότι για την υπόθεση του 8% η Κομισιόν ήταν ξεκάθαρη και Ακούω τα όσα λένε οι διαπραγματευτέ από νομική και πολιτική φύση για τη σαφή φύση σε επίπεδο 1, αυτό το 8% να εξεταστεί αναπερίπτωση περίπτωση και να μην αποτελεί τον κανόνα. Ίσως όμως θα έπρεπε να ρωτήσουμε την Κομισιόν πώς, και συνδέεται, πώς μάλλον δεσμεύουν όλα αυτά το Συμβούλιο. Γιατί εμεί είμαστε συνομοθέτες τρίτη, ε, τρίτο θέμα το οποίο ε, δεν λέγεται ποτέ ρητά, αλλά εννοείται ε, είναι να ρωτήσουμε την Κομισιόν μήπως μία από τις δυσκολίες που έχουμε δεν σχετίζεται με το θέμα του ότι η μία ε, εξυγίανση δεν βασίζεται σε προηγούμενες ε, ρυθμίσεις, γιατί όλα έχουν γραφτεί, λες και υπέρχει επιλογή ανάμεσα ε, σε κάτι, όμως η εξυγίανση είναι κάτι, είναι μια πολιτική λύση πολύ πιο δαπανηρή από αυτή που αρχικά έχει προβλέψει ο νομοθέτης. Αυτό έχει να κάνει με ψυχολογία, πολιτική κτλ. Πράγματα που δεν μπορούμε να αποσιωτικοποιήσουμε, αλλά που επηρεάζουν τη συζήτησή μας όσον αφορά την εφαρμογή του 8%. Πώς λοιπόν θα κάνουμε σε σχέση με αυτό το κίνδυνο που κατά τη γνώμη μου δεν ελήφθη υπόψη στη φάση της σύνταξης της νομοθεσίας. Γιατί είπαμε όταν το κάναμε αυτό, ναι, θα υπάρχουν τράπεζες που θα πρέπει να εξηγηθούν, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν είδαμε πώς. Στην πράξη όμως, στην πολιτική, βλέπουμε ότι αυτή η εξηγήνση εξαιρετικός καθίσατε δυνατή. Thank you, Sven Giegold. Sven Giegold. Thank you. First, uh, Σας ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την Ελίζα για την καλή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα και αν ποτέ δεν συμφωνούσαμε 100% και ιδιαίτερα σε τούτο εδώ το θέμα, αλλά εκτιμώ όλα αυτά τα χρόνια την εμπιστοσύνη και την αγαστή συνεργασία που είχαμε. Και επίσης να καλωσορίσω και την Περβάνς Περές ως νέα συντονίστρια για τους συντονιστές από πλευρά των Πρασίμων και είμαι βέβαιος ότι αυτό το πνεύμα συνεργασίας που πάντοτε ε, διέπνε όλα τα κόμματα σε αυτή την εδώ την Επιτροπή θα συνεχίσει να ισχύει. Και σου εύχομαι καλή τύχη στην Πορτογαλία, στην Κεντρική Τράπεζα Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Και φυσικά καλωσορίζω το γεγονός ότι μετακινήσεις σε ένα δημόσιο αξίωμα παρά να μετακινηθείς σε ένα λόμπι. Σε ευχαριστώ λοιπόν που εξακολουθείς να στηρίζεις το κοινό καλό για το δημόσιο τομέα. Σε ευχαριστώ. Ε, εδώ τώρα όμως ε, θέλω να πω κάποια ξεκάθαρα πράγματα και θέλω μαζί σας να πω ότι αυτό το θέμα το θεωρώ πολύ συμβολικό που δείχνει δηλαδή την ευρύτερη εικόνα. Το Κοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση BALTS, που είναι μια ισορροπημένη συμβιβαστική για το τι θα κάνουμε τώρα με την κατάσταση της νομοθετικής μας, ε, της, ε, συγγνώμη, χρηματοπιστωτικής μας νομοθεσίας. Εντάξει, μετά από μια τόσο βιαστική μεταρρύθμιση, τίποτα δεν είναι τέλειο, το ξέραμε αυτό. Αλλά ζητάμε όχι να αποδυναμωθεί η νομοθεσία, αλλά να ενισχυθεί σε κάποιους τομείς, να διορθωθεί κάπου αλλού, να αναζητηθούν τα κενά καθώς και τα σημάδια επιβα... υπερβολικής επιβάρυνσης κτλ. Ήταν ισορροπημένη αυτή η θέση. Βλέπουμε λοιπόν τι συμβαίνει τώρα και τα διάφορα στάδια του ίδιου διάφορα μάλλον σκηνικά του ίδιου θεατρικού έργου. Βλέπουμε συστηματικά να, επιχειρούνται, να επιχειρείται η αποδυνάμωση και με σοκάρισε η διάσκεψη της Κομισιόν μετά από τη διαβούλευση στην οποία συμβάλαμε και εμείς. Γιατί για μένα αυτό δεν ήταν ισορροπημένη συμβιβαστική αυτό που παρουσίασε η Κομισιόν ως προτάσεις μετά από αυτήν την ε, διαβούλευση. Αλλά ένα ευχολόγιο πολύ μονομερές. Και τώρα όσον αφορά τις τράπεζες βεβαίως αυτό το ανέφεραν και διάφοροι ομιλητές Ξέρουμε ότι στο Συμβούλιο δεν πιστεύουν όλοι σε αυτό που αποφασίσαμε και όχι στην τελειοποίηση, δεν λέω για τις λεπτομέρειες, αλλά για τα βασικά στοιχεία. Το bail-in, ισχυρές κεφαλαϊκές απαιτήσει είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε σε μια οικονομία χωράς με ιδιωτικέ τράπεζες και πιστεύουμε ότι εφόσον έχουμε ιδιωτικέ τράπεζε μετά και από αυτή την κρίση, ε, υπάρχουν ε, λόγοι στου οποίου οφείλεται αυτό και πρέπει να μπορούν να φέρουν του κινδύνου του, τα ρίσκα ίδιε. Γιατί πρακτικά, γιατί να έχουμε οικονομία τη αγορά. Και υπάρχουν διάφορα στάδια τώρα όπου διάφορα κρατημέλη ζήτησαν την αποδυνάμωση των στάνταρ. Έχουμε λοιπόν σαφή δέσμευση από διάφορους βασικούς παίκτες ε, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Εξυγίανσης και τη Κομισιόν για ελάχιστες απαιτήσει για πρόσβαση στο Ταμείο. Το λογικό συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο έμρελ, γιατί διαφορετικά δεν είναι λογική η κατάσταση. Και τώρα μαθαίνουμε ότι κράτη-μέλη, Ιταλία και Γαλλία στο Συμβούλιο πιέζουν να είναι αναπερίπτωση η μεταχείριση και το 8% είναι εξαίρεση και όχι το μίνιμουμ και ότι η Κομισιόν υποχώρησε και στήριξε αυτή τη θέση μέσω αυτή τη στενή και πολιτική ερμηνεία αυτή τη προδιαγραφή που είναι τώρα υποσυζήτηση. Οπότε το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο. Θα είναι μέρος του απόπειρα να αποδυναμωθεί η κατάσταση και να ακολουθηθεί το ευχολόγιο ορισμένων φορέων ή θα κρατήσουμε σταθερή θέση και το 8% κεφαλαικών απαιτήσεων θα καταστεί το μίνιμουμ για να μπορεί με ασφάλεια να λειτουργεί μια ιδιωτική τράπεζα στην κοινή αγορά. Αυτό είναι το ερώτημα και δεν θα πρέπει να βάλουμε τρικλοποδιά στο Συμβούλιο Εξυγίανσης, αλλά να το στηρίξουμε με συγκεκριμένα και σαφή μηνύματα, ώστε να πείσει τα κρατημέλη να θεσπίσουν το 8% ως ελάχιστο όριο. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, Σβέν. Έχω και εγώ κάποιες ε, ερωτήσεις. Ε, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες ε, ερωτήσεις, γιατί θέλω να σας πω ότι δεν συμφωνώ με την ανάλυση σας, αυτό είναι απόλυτα σαφές, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή και ο κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτή η συζήτηση. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Η μία φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη δουλειά της για το ΤΙΛΑΚ και πώς ακριβώς εξετάζεται το θέμα του εύρους του ΤΙΛΑΚ. Υπάρχει το θέμα των e και G-SIPS. Δεύτερον, έχω μία ερώτηση για την Ελκε König γιατί έχω το κείμενο της ομιλίας σας και είπατε ότι η SRB δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αλλάξει πολιτική ως αποτέλεσμα αυτής της κατεξουσιοδότηση πράξης. Φαντάζομαι αναφέρεστε στο ότι αφού έχει περάσει η περίοδος ελέγχου, αυτή η πράξη γίνεται νόμιμη πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ακριβώς εννοείται με αυτό που λέτε, ότι η ε, πράξη πρέπει να είναι συνεπής ή να είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια διευκρίνηση. Γιατί κατά την άποψή μου η κατεξοδότηση πράξη είναι ένα τμήμα της νομοθεσίας που λέει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται τα άρθρα 42.6 και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όλοι οι θεσμοί να ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο το νομικό κείμενο και να το εφαρμόζουν και με συνεπή τρόπο. Κατόπιν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε ότι ΕΜΡΕΛ πάνω από 8% ε, θα αφορούν τις μεγάλες τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι είπατε, αλλά δεν το κατάλαβα καλά. Τι ακριβώς εννοείτε με τις ε, μεγαλύτερες τράπεζες, της g ή όλες τις ε, τράπεζες υπό την ομπρέλα του νέου, νέου Συμβουλίου Εξυγίανσης, και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Γιατί βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τροποποιεί μία κατεξοδότηση πράξη της ε, Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Αρχής και τροποποιεί και ένα άρθρο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες. Και τέλος, όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες, στην ε, Ευρωζώνη και γενικότερα. Αυτή είναι μία ερώτηση προς όλους τους θεσμούς, γιατί τα δύο εργαλεία είναι διαφορετικά. Ε, όταν το TILAC είναι πιο ήπιο, τα, DEMIREL, τα MREL είναι πιο σκληρά και ε, αν δούμε την νομική ευθύνη, βεβαίως και βλέπουμε ότι διαφέρουν όλα αυτά. Ε, στο δεύτερο πυλώνα, αν δούμε λιγάκι το πρόσφατο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό που έχει σημασία είναι σε τελική ανάλυση ε, πώς μπορούμε να έχουμε ένα συνεπή, ε, ευανάγνωστο μηχανισμό, όχι απλά την επικάλυψη διαφορετικών κριτηρίων. Θέλω λοιπόν να γνωρίζω πώς πιστεύετε ότι αυτά τα MREL και τα TLAC πώς ε, πρέπει να τα εντάξουμε στην νομοθεσία μας και κατά πόσον όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στο να έχουμε ένα εξορθολογισμένο ευανάγνωστο μηχανισμό για να διαχειριστούμε τη σταθερότητα αλλά και τις ίσες ευκαιρίες. Αυτή έτσι είναι μια γενικότερη ερώτηση που σας υποβάλλω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σημαντικά τα ερωτήματα. Θα ξεκινήσω με αυτό που είπε ο κύριος Χέκμαρκο, εισηγητής, για να μην υπάρχει παρανόηση. Εμείς πιστεύουμε ότι το πρώτο που προτείνει η EBA θα μπορούσε να ακυρωθεί από το δικαστήριο. Είναι νομική πράξη της Κομισιόν το κείμενο. Τώρα, κάτι πολύ σημαντικό για την ουσία. Για να μην υπάρχει παρανόηση δύο πραγμάτων, μεταξύ δύο πραγμάτων. Κατώτατο ποσοστό 8% MREL και κατώτατο 8% bail-in πέντε στο ταμείο. Ίσως εκεί υπάρχει κάποια παρανόηση. Θέλω λοιπόν να είναι ξεκάθαρο και για να μην υπάρχει λοιπόν παρανόηση, επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνει αλλαγή στο κανόνα 8% ε, Μπέιλιν. Ε, Πριν υπάρχει πρόσβαση. Να μην προτείνει μάλλον κάτι τέτοιο το Κοινοβούλιο, γιατί δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα στο τραπέζι. Το 8% έμρελ, κατώτατο ποσοστό. Στη μελέτη αντικτύπου, ναι, κάνουμε, ξέρετε, στην Κομισιόν, ίσως όχι για τα πάντα, αλλά κάνουμε μελέτη αντικτύπου. Λοιπόν, εκεί για την οδηγία, την ανάκαμψη και την εξυγίανση, λέμε ότι από τις 30 υποθέσεις που εξετάσαμε, τρει μόνο χρειαζόταν απορρόφηση ζημιών και ανακεφαλαιοποίηση ποσοστού πάνω από 8 MRL. Δεν είναι ο μαγικό άριθμο αυτό, απλά για να ξεκαθαρίσω αυτό που είπε η κυρία Φερέιρα. Το κατώτατο αυτό ποσοστό 8% έμρελ θα πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα και στην πραγματικότητα. Μέχρι στιγμή δεν είχαμε τέτοια δεδομένα, δεν είχαμε τέτοια εμπειρία μέχρι τώρα και γι' αυτό πιστεύουν ότι η αρχή εξυγίανση και το Συμβούλιο Εξυγίανση, SRB θα πρέπει να έχουν την ευελιξία, αλλά τράπεζα να εφαρμόζουν αυτό που θεωρούν ε, σκόπιμο. Διαφορά λοιπόν μεταξύ 8% Μπέιλιν, αυτό δεν ε, συζητείται, 8% MRL είναι κάτι διαφορετικό. Χρειαζόμαστε ευελιξία για τις αρχές εξυγίανσης. Ο ε, κύριος Μπάλτς έθεσε σημαντικά ερωτήματα, 3,5% ε, είναι κάτι που το πολεμήσαμε για το FSB και ως Κομισιόν και θέλουμε να υλοποιηθεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, να το περιμένετε. Επίσης και η απαιτήση για τον πυλώνα 2 είναι πολύ σημαντικά κύριε Μπάλτς. Θα το θα το δείτε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι το οποίο είπε η κυρία Γκουλάρ. Εδώ είμαι, έχω αλλάξει θέση. Πίσω. Α, σας έψαχνα, γιατί εξαφανιστήκατε ως διαμαγείας. Λοιπόν, είναι από το EFSB αυτή η πρόταση. Δεν ε, έχει την ισχύ ε, ενωσιακού δικαίου. Γι' αυτό και έχουμε υποβάλει πρόταση για ένα ενωσιακό νομοθέτημα, ώστε κοινοβούλιο και συμβούλιο νομοθέτε να νομοθετήσουν, να εγκρίνουν το σχετικό νομοθέτημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό από πλευρά δημοκρατίας. Δηλαδή, πρόταση και θα έχει προηγηθεί πλήρης ε, ανάλυση αντικτύπου από την Κομισιόν ως ήθιστε. Επόμενο σημείο, αυτό που είπε η κυρία Μπερές για το ε, το χρειαζόμαστε τώρα, τα είπε η κυρία Κένικ. Το TILAC το χρειαζόμαστε ε, το 2017. Δύο δεσμεύσεις που νομίζω ότι μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Ελπίζω να έχω τις περισσότερες ε, ερωτήσεις και σας δώσω συγγνώμη αν μακρηγόρησα. E Ευχαριστώ η EBA, Ευρωπαϊκή Αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, για το 8%. Το βασικό που θέλω να τονίσω, το είπε και η Κομισιόν, και από το SRB, δεν περιμένουμε οι τροποποιήσει τη Κομισιόν να αλλάξουν ε, την πολιτική για τα MRL που εγκρίθηκαν από τις αρχές εξυγίανσης. Ε, το SRB λέει ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει η πολιτική και αυτό συνάδει και με το πώ εμεί αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση και από άλλες αρχές εξυγίανση εκτό Ένωση που έτσι έχουν προχωρήσει αν έχουν πολιτική δηλαδή συγκεκριμένη για το θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο του FSB, είπε και η Κομισιόν, η εντολή μας ε, μας δίνεται από τους νομοθέτες και όχι από το FSB. Πολλά ε, μέλη μας φυσικά συμμετέχουν συζητήσεις του FSB και μας μεταφέρουν και αυτή την προοπτική. Όμως η νομοθετική μας εντολή προέρχεται και το λέω ξεκάθαρα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ορισμένοι ανέφεραν τη συμβατότητα μεταξύ TLAC και ΕΜΡΕΛ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι ενιαία και συνεκτική η δέσμη των απαιτήσεων αν έχουν να επιτύχουν τους ίδιους στόχους, γιατί θα ήταν δύσκολο ε, για τις τράπεζες. Να έχουν δύο διαφορετικές δέσμες απαιτήσεων με διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές, ίδιους στόχους όμως. Και επίσης θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να είναι ισότιμο το πεδίο ανταγωνισμού με αναλογική εφαρμογή των MRL. Και τέλος, πολλοί ρώτησαν μπορεί να προστευτεί το πλαίσιο. Νομίζω ότι ναι. Θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιες ευκαιρίες όταν θα εφαρμόσουμε τα, το TILAC. Ίσως στην περίπτωση των τεχνικών προτύπων. Θα μπορούσαμε, αν στο επίπεδο 1 έχουμε κάποιες αλλαγές, να ε, εποφεληθούμε αυτής της δυνατότητας. Όταν βέβαια έχει ολοκληρωθεί και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ, Ελκε Κένικ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να επαναλάβω μία πρόταση και μετά θα πω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε ο Πάτρικ Πίρσον και ο πρόσωπος της EBA. Ε Τα MRL είναι το βασικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή του οι αρχέ εξυγίανση για να πετύχουν την δυνατότητα εξυγίανση των τραπεζών. Συμφωνώ επομένω και πιστεύω απόλυτα ότι αυτό είναι ο σωστό τρόπο να προχωρήσουμε. Δεν είναι δηλαδή αποφάσεις που λαμβάνονται ανά τράπεζα, αλλά από το συστημικό αποτύπωμα εξαρτάται. Από το συστημικό αποτύπωμα των τραπεζών. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αρχές εξηγήσεις να έχουν τη δυνατότητα και την εξουσία να ορίζουν τα MRL για να πετύχουν αυτό το στόχο της δυνατότητας της ε, γιατί λέτε, εμείς δεν βλέπουμε ανάγκη να αλλάξουμε την πολιτική μας. Το συζητήσαμε διαμακρών. Κατά πόσον δηλαδή διαγραφή του 8% και αυτή η τετραετία ε, συνιστά μείζωνα αλλαγή ή όχι. Εμείς βασίσαμε την πολιτική μας ε, στο σχέδιο ε, του, της CBA. Όταν μιλάμε για 8%, και εδώ έρχομαι στο δεύτερο σας ερώτημα. Εστιάζουμε ξεκάθαρα στις τράπεζες που είναι στο, στο πεδίο εντολή ε- του, του, του, του, Συμβουλίου Εξυγίανσης. Αλλά βέβαια αυτό το μπορεί να υπερβαίνει πολύ αυτό που θα χρειαστεί κάποια τράπεζα. Υπάρχουν όμω κάποιε τράπεζε που για την Ένωση ή για το μεμονωμένο κράτο μέλο, το εκάστοτε, είναι οι σημαντικότερε τράπεζε. Και αν δείτε και το όλο οποίο, έχετε τι G-SIPs. Κάποιε από τι ε, G-SIPs που δεν έχουν στην Ευρωζώνη είναι πολύ λιγότερο σημαντικέ στην Ευρωζώνη σε σχέση με κάποιε άλλε τράπεζε που δεν είναι G-SIP. Δεύτερη-τρίτη γραμμή τράπεζε και ούτω καθεξής. Άρα για εμάς σημαντικό είναι ποιες τράπεζες θα χρειαστούν αυτό το 8% αποδεκτών υποχρεώσεων bail-in. Συμφωνήσαμε ε, και είπαμε λοιπόν ότι ίσως καλό θα ήταν και λογικό να έχουμε και ένα 8% MRL ως αρχή. Τέλος, ισότιμο του ανταγωνισμού. Γιατί. Βλέπουμε και τι κάνουν άλλες αρχές εξυγίανσης. Έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τραπεζών στην Ευρωζώνη, αλλά και σε σχέση με άλλα κράτη μέλη. Βλέπουμε τα TILAC, τα EMREL και προσπαθούμε ε, να πετύχουμε τον στόχο ε, του να είναι οι τράπεζες δυνατόν να εξυγιανθούν Τώρα αν θα υπάρξει παγωγή, αν θα δούμε πού θα βάλουμε το MRL σε σχέση με το TILAC. Αλλά πάντα μιλώ για τις πιο μεγάλες τράπεζες. Υπάρχουν και πιο μικρές τράπεζες όπου το μηδέν ή λίγο παραπάνω είναι μια χαρά, αλλά για τις μεγαλύτερες τράπεζες μιλάμε. Αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και όταν θα καθορίσουμε τα MRL. Για μας το είπα ξεκάθαρα. η η κανονισμή οδηγία για ανάκαμψη τα λοιπά είναι το πλαίσιο. Όλα τα άλλα είναι ιδέες, το τα εξετάσουμε. Αλλά πάντα στο νομικό αυτό πλαίσιο που κινούμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς ε, πολύ. Ευχαριστούμε όλους όσοι έλαβαν το λόγο για τη συνεισφορά του στη συζήτηση. Και ε, θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης ε, θα συζητήσει, θα τοποθετηθεί για την κατεξοδότηση πράξη δεν ξέρω αν κύριε Σιγητά θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, εγώ νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πρέπει να βυθιστούμε περισσότερο σε όλα αυτά τα ερωτήματα, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές διαφορές. Αλλά πραγματικά μου άρεσε πολύ η συζήτηση και ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Άρα κλείνει αυτό το σημείο της σημερινής διάταξης και πάμε στο επόμενο θέμα που είναι ο διορισμός του Προέδρου της ΕΦΡΑΚ. Και θα ήθελα να, καθορίσω, να καλωσορίσω τον Ζαν Πολ Γκοζές. Χαιρόμαστε Ζαν Πολ που σε έχουμε κοντά μας στην Επιτροπή όπου παίξατε πολύ σημαντικό ρόλο για πάρα πολλά χρόνια και όπως πολύ καλά γνωρίζετε Ο κύριος Γκοζές ε, είναι ο υποψήφιος που η Κομισιόν πρότεινε για την θέση του Προέδρου της ΕΦΡΑΚ. Και με βάση τους ε, κανόνες πρέπει τώρα να κάνουμε ακρόαση με τον κύριο Γκοζές και θα ψηφίσουμε σήμερα για το διορισμό του. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, καλωσορίσω και σας δίνω ευθύς αμέσως ε, το λόγο για την ομιλία σας ε, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τις ερωτήσεις από τα μέλη μας. Ζαν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κατανοήσω ότι με μια κάποια συγκίνηση βρίσκομαι πάλι εδώ σε αυτή την αίθουσα και βλέπω ε, γνωστά και φιλικά πρόσωπα. Η μοίρα ε, οδηγεί, αφού πέρασα 10 χρόνια εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, 10 χρόνια στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, μετά από 2 χρόνια αναμονής ε, τόλμησα να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία της ΕΦΡΑΚ. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η υποψηφιότητα είναι λίγο είναι λίγο φιλόδοξη, γιατί δεν έχω τις γνώσεις και την εμπειρία του προκατόχου μου, αλλά ελπίζω με τη δική σας εμπιστοσύνη να μπορέσω να σταθώ σε αυτή τη θέση. Η οικονομική και η νομική μου ε, μόρφωση να βοηθούν. Ήμουν πολύ γρήγορα βοηθός στο Πανεπιστήμιο που δίδαξα ε, ε, πολιτική οικονομία και δίκαιο. Ε, ε, στη συνέχεια για 15 χρόνια δούλεψα ως νομικός στο Συμβούλιο Επικρατείας και τέλος επαγγελματική μου σταδιοδρομία ήταν ότι ήμουν νομικός και οικονομικός διευθυντής μιας τράπεζας που είχε ειδικευθεί στη χρηματοδότηση τοπικών συνεταιρισμών. Διέκοψα την επαγγελματική μου δραστηριότητα για να αφιερωθώ αποκλειστικά στην ε, θητεία μου ως Ευρωβουλευτή και επίσης εγκατέλειψα τις τοπικές μου αρμοδιότητες γιατί 30 χρόνια διατέλεσα δήμαρχος μιας μικρής κοινότητας 300 κατοίκων. Εκτός της Γαλλίας αυτό κάνει τους άλλους να γελούν γιατί στη Γαλλία έχουμε πολύ μικρούς δήμους και κοινότητες. Ήμουν λοιπόν δήμαρχος μιας μικρής κοινότητας της Νορμανδίας για 30 χρόνια. Στο Ευρωκοινοβούλιο, οι συνάδελφοι που είναι εδώ το γνωρίζουν, ότι είχα την τιμή να είμαι συντονιστής της ομάδας του ΕΛΚΑ από το 2007 μέχρι το 2014 και συνεργάστηκα με τον φίλο Μπάλτς. Συμμετείχα στην επεξεργασία διαφόρων σημαντικών θεμάτων όπως την οδηγία EFMB, τους πρώτους κανονισμούς ε, για τους οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας και τα λοιπά, αλλά είναι σαφές ότι τα προσόντα που ζητώνται για τον έφραγ είναι ευρύτερα. Ωστόσο, η εφράγα αναδιοργανώθηκε μετά από την έκθεση του, του Φίλιπ ε, Μέστατ και η θέση του Προέδρου της ΕΦΡΑΓ είναι κάπως παράξενη. Δηλαδή, αν δούμε το καθεστώς, ε, το καταστατικό δεν βλέπουμε μεγάλη ακρίβεια για το τι κάνει, ωστόσο πρέπει να έχει ένα ρόλο συνδετικό αλλά και να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον, διότι μία από τις ιδιαιτερότητες της ΕΦΡΑΓ είναι να αποτελείται ταυτόχρονα από τους stakeholders, ε, τους ενδιαφερόμενους φορείς που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα συμφέροντα, τους ρυθμιστές των διαφόρων χωρών και τον πρόεδρο, ο οποίος δεν είναι ούτε από τη μια μεριά ούτε από την άλλη. Και τέλει, ίσως και αυτή να είναι η καινοτομία στο project αυτό που ετέθησε σε εφαρμογή μετά από τις συστάσεις του κυρίου Μέστεγ. Δεν χρειάζεται να σας πω για τους κανόνες που είναι υπό εξέταση, γιατί η ΕΦΡΑ γνωρίζεται ότι αποτελείται από διάφορα επίπεδα, έχει μια επιτροπή τεχνική, ε, ιδιαίτερα ειδικευμένη, ένα συμβούλιο και έχει και ένα αρμόδιο τεχνικά προσωπικό για αυτά τα πολύ ειδικά θέματα. Να σας πω περισσότερο πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τη δράση του Προέδρου του ΕΦΡΑΓ. Σε αυτή τη νέα οργάνωση θα πρέπει να μεριμνήσω τα διάφορα επίπεδα αρμοδιοτήτων να λειτουργούν αρμονικά και να εφαρμόσουμε μαζί με τον Διευθυντή, γιατί υπάρχει ένας Γενικός Διευθυντής που έχει την ευθύνη για το προσωπικό, να θέσουμε σε εφαρμογή τις διατάξεις που θα επιτρέψουν στην ΕΦΡΑΚ να παίξει πλήρως το ρόλο της στο συμβουλευτικό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση, τη διαπραγμάτευση των διεθνών λογιστικών κανόνων. Και όταν λέω να παίξει πλήρως το ρόλο της, το λέω διότι το τι έχει γίνει μέχρι τώρα είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούμε να τα πάμε και καλύτερα έτσι ώστε η φωνή της Ευρώπης να είναι ισχυρότερη στην εφαρμογή της ε, ε, τυποποίησης ε, της λογιστικής διεθνώς. Η Ευρώπη επέλεξε να μην έχει ένα δικό της τύπο, αλλά να δεχτεί τους κανόνες που επεξεργάζεται η Διεθνής Ομοσπονδία, η πέρα από το καταστατικό αυτού του οργανισμού. Και τώρα η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με τη δική της φωνή έτσι ώστε η τυποποίηση που ετοιμάζεται να είναι συμβατή και σύμμορφη με τις αρχές που διέπουν την λογιστική πολιτική στην Ευρώπη όπως η πιστή απεικόνηση, η φρόνηση, η αξιοπιστία αλλά οι κανόνες αυτοί να λαμβάνουν υπόψη και τις ειδικέ ανάγκες της Ευρώπης. Και κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο ρόλος του Προέδρου να μεριμνήσει ώστε οι κατευθύνσεις αυτές τις γραμμές να είναι πραγματικά, να εφαρμοστούν πραγματικά. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι οι μελέτες αντικτύπου που υπάρχουν και που είναι ήδη ικανοποιητικέ να λαμβάνουν υπόψη περισσότερο τις μακροοικονομικές συνέπειες της έγκρισης των κανόνων με τρόπο ώστε οι συνέπειες αυτής της ε, λογιστικής μεθόδου στην οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική σταθερότητα είδαμε ότι ορισμένες ταξινομήσεις, ορισμένες χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν επιταχυντές της κρίσης αντί να αποτελέσουν σταθεροποιητικά στοιχεία. Αυτές είναι κάποιες συγκεκριμένες δράσεις λοιπόν ενέργειες, τις οποίες θα πρέπει να προβεί ο πρόεδρος της ΕΦΡΑ και θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το δημόσιο συμφέρον. Ο Φίλιπ Μέστα στη δική του έκθεση άρχισε να εκπονεί, να επεξεργάζεται κάποια στοιχεία αυτού του τύπου. Θα πρέπει βεβαίως να εμβαθύνουμε στα κριτήρια και να διαπιστώσουμε για να τα αντροποποιήσουμε δεχομένως τι συνέπειες έχουν οι το η... η λήψη υπόψη του δημοσίου συμφέροντος στους ε, κανόνες, στους λογιστικούς. Αλλά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον, ένα εταίρο είναι απαραίτητο. Είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Παλιότερα το Κοινοβούλιο θα έλεγα ότι ήθελε να βελτιώσει και να ενισχύσει τους κανο... τους τις σχέσεις με τους τρεις οργανισμούς Νομίζω όμως πως μια εναρμόνιση με τους οργανισμούς αυτούς είναι σημαντική έτσι ώστε η αναζήτηση της ε, συνένεσης που είναι απαραίτητη ώστε να έχουμε φωνή διεθνώς να γίνει και στην πραγματικότητα. Οι θέσει που είχα εδώ σε αυτή την επιτροπή μου είχαν δώσει την ευκαιρία να έχω προσωπική επαφή με τους τρεις προέδρους των οργανισμών και ελπίζω να εκμεταλλευτώ αυτή την καλή μου σχέση ώστε να Ε, λειτουργεί πιο αγαστά η συνεργασία ανάμεσα σε όλους αυτούς τους οργανισμούς. Και όσο για το Ευρωκοινοβούλιο, διάβασα με πολύ ενδιαφέρον την έκθεση που έφτιαξε ο Θεοδόρος Τόλογεν, την οποία ψηφίσατε και που θα περάσει από την Ολομέλεια τον Ιούνιο και όπου περιλαμβάνονται πολλές παρατηρήσεις που είναι πολύ κέρυες, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πάντως εγώ θα τις χρησιμοποιήσω αν μου εμπιστευτείτε αυτή τη θέση. Θα ήθελα λοιπόν να σας δηλώσω σαφώς ότι επιθυμώ και δεν είναι απλώς επιθυμία, είναι επιθυμία του θεσμού. Θα ήθελα να έχω με το Κοινοβούλιο περισσότερο από ό,τι παλιά σχέσεις εμπιστοσύνης και σχέσεις ε, στενή συζήτηση. Δηλαδή, να μπορούμε να διοργανώνουμε από καιρού καιρών, είτε μετά από αίτημα της ΕΦΡΑΚ, είτε μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου, και μάλιστα του Πρόεδρου της ομάδας που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε όσους παρακολουθούν πιο συγκεκριμένα τα λίγο περίπλοκα και, ε, και κομμάτια και θέματα, να μπορούμε να συζητήσουμε λοιπόν για το τι θα πρέπει να έρθει επιτάπητος, γιατί η δεν μπορεί μόνο να αντιδρά, θα πρέπει να είναι και να είναι ναι, αλλά να είναι και δραστήρια. Να θίγει ζητήματα πριν να τα σκεφτούν άλλοι. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, βαρύνουμε με την παρουσία μας, όχι να περιμένουμε κατόπιν εορτής να υποβάλουμε συστάσεις. Η και συμβουλεύει την, την Επιτροπή, αλλά εγώ είμαι πιο πολύ συνδεδεμένος με το Ευρωκοινοβούλιο και είμαι έτοιμος και πολύ γρήγορα όταν και αν αναλάβω αυτή τη θέση, να κάνουμε μια πρώτη σύνοδο εργασία ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους ευρωβουλευτές, ώστε να Έχουμε στενές συναδελφικές σχέσεις. Ως συντονιστή, έχω την, την, την συνήθεια να συνεργάζομαι με συναδέλφους όλων των ομάδων, προσπαθώντας να βρω ευφυείς ε, λύσεις και ε, συμβιβαστικέ ε, λύσεις. Έτσι δεν υπάρχει σε αυτή τη συναδελφική εργασία να μην γίνει και σε αυτό το πλαίσιο στη σχέση δηλαδή με το Ευρωκοινοβούλιο. Ε, είμαι στη διαθέσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις που ελπίζω να μην είναι πολύ δύσκολες. Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική, να πω, παρουσίαση που υπόσχεται και πολλά σε σχέση με τις ε, επαφές μας και τον ε, ενεργητικό ρόλο της ΕΦΡΑΚ. Να περάσω στους ε, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Γύρω στα 3-4 λεπτά να διαθέσουμε, γιατί έχουμε και ψηφοφορία, κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ζαν Πολ. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ομολογήσω ότι σήμερα σε μια τέτοια κρόαση δεν μπορώ να είμαι ε, τελείως ουδέτερος λόγω της ε, μακροχρόνιας ε, φιλίας μας και γιατί συνεργαστήκαμε και τόσο καλά. Βλέπει κανείς πόσο καλά γνωριζόμαστε από το γεγονός ότι τα ερωτήματα που έχω σημειώσει ήδη καλύφθηκαν από αυτά που μας είπες. Βεβαίως αυτό που μου άρεσε καλύτερα ήταν αυτό που είπες για τη σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που εντάξει το θεωρούσα και λιγάκι αυτονόητο. Για μένα υπάρχει άλλο ένα ερώτημα, επειδή το ανέφερες ε, πολύ συνοπτικά λόγω του περιορισμένου χρόνου. Είπες ότι η Ευρώπη οφείλει να εκφράζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ακόμα και σε θέματα ε, διεθνούς βεληνικούς, ανταγωνισμού ή οτιδήποτε. Μήπως μπορείς λιγάκι να το διευκρινίσεις αυτό, γιατί για μένα αυτό είναι ένα από τα βασικότερα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν κατά τα επόμενα έτη. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε σήμερα κοντά μας ως υποψήφιος και νομίζω αυτό δεν ισχύει μόνο για μένα προσωπικά, αλλά για το σύνολο της ομάδας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. είπα ότι ότι η ΕΦΡΑΚ με τις ε, τεχνικές σχέσεις που θα έχει θα ε, είναι πιο δυνατή με την έννοια ότι θα είναι για τις διάφορες ευρωπαϊκές θέσεις με στόχο τη δημιουργία μιας ισχύρης ε, συνένεσης και θα ήταν πιστεύω επιζήμιο για την Ευρώπη η ΕΦΡΑΚ να δίνει στην Κομισιόν κάποιες συμβουλές που θα τις ακολουθήσει, θα τις ακολουθήσει και παράλληλα στην Ευρώπη να δίνονται τελείως διαφορετικές απόψεις για σημαντικά ζητήματα. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε όλη η ομάδα της ΕΦΡΑΚ, ώστε να έχουμε την όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση για τις θέσεις τις οποίες ε, λαμβάνουμε σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ενεργητικοί, εκ των προτέρων να προδικάζουμε κάποιες συζητήσεις, να αποκαταλαμβάνουμε δε, ενδεχομένως και κάποιες αντιφάσεις ή διαφορές που θα ήταν επιβλαβείς για την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι σημαντική δουλειά που έχουμε να κάνουμε και με βάση όσα γνωρίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να μας δώσει βαρύτητα Γι' αυτό και η ΕΦΡΑΚ τροποποιήθηκε εν μέρη, χωρίς αυτό βέβαια να αμφισβητεί το τι έκανε μέχρι τώρα και το πώς λειτουργήσαν μέχρι τώρα οι ομάδες της. Επιμένω επίσης στο γεγονός ότι πρόεδρος και γενικός διευθυντής θα πρέπει να εργάζονται σε απόλυτη αρμονία. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός εξουσίας. Σήμερα το πρωί μίλησα στο τηλέφωνο του Γενικό Διευθυντή. Άγγλος είναι και αγγλόφωνος. Και του είπα, η μόνη ε, μας ανταγωνισμός που υπάρχει ε, μεταξύ μας είναι ποιος μιλάει πιο καλά τη γλώσσα του άλλου. Έτσι, για να πω και ένα αστείο. Η ΕΦΡΑΚ πρέπει να είναι ένα μπλοκ ενωμένο που ε, θα το διευθύνουν με αρμονία ε, το δίδυμο των προέδρων και, του Γενικού Διευθυντή. Κύριε Μπερέ, σε ευχαριστώ. Ζαν Πολ, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Είμαι και συντονίστρια της ομάδας Σοσιαλιστών Δημοκρατών νέο ε, καθήκον. Ξέρω ότι εσείς το έχετε επιτελέσει με, απόλυτο, με απόλυτη επιτυχία κατά το παρελθόν. Τρεις ερωτήσεις έχω. Καταρχάς, την έφρακτη γνωρίζουμε εδώ και καιρό αρχικά την είχαν πλασάρει όπως εσείς την περιγράφετε τώρα ότι είναι ο συνήγορος ε, της Ευρωπαϊκής Οδού. Πολλές φορές είδα όμως να γίνεται το αντίθετο η ΕΦΡΑΚ. δηλαδή να είναι η δικηγόρος του ESB στην Ευρώπη και όχι το αντίστροφο. Πώς θα εφαρμοστούν λοιπόν αυτά που επιθυμεί ο Φιλιπ Μέιστα. Δεύτερον, για την διαδικασία ορισμού. Και για την περίοδο αυτή, ε, τη μεταβατική, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό επηρεάζει τη λειτουργία του θεσμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενδεχομένως. Επίσης, λέτε ότι θέλετε να λάβετε υπόψη τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Υπάρχει ένα επίγον καυτό θέμα στην επικαιρότητα, το IFRS e 9. Πολλοί Ευρωπαίοι διερωτώνται για αυτά τα πρότυπα χρηματοοικονομική πληροφόρηση πώ θα υποστηρίξουν τι μακροχρόνιε επενδύσει. Πιστεύετε ότι η συνθήκη που παρενέβη τελικά η ΕΦΡΑΚ σε αυτή την αξιολόγηση είχε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τη ή θα πρέπει να βελτιώσουμε τις μελέτε αντικτύπου, για την εφαρμογή ενό λογιστικού προτύπου. Έχω και άλλα ερωτήματα, αλλά θα σα δώσω το λόγο να απαντήσετε, γιατί αλλιώ δεν θα είναι εύκολο. Πάντω, ναι, και αυτά ήδη ήταν δύσκολα ερωτήματα. Ο κ. Γκοζές, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, γιατί για μένα παραμένετε πρόεδρο τη Επιτροπή ΕΚΟΝ από την πρώτη μου θητεία. Σα ευχαριστώ λοιπόν για αυτέ τι ερωτήσει. Σε ό,τι αφορά τι σχέσει ε, με το ΡΙΑΣΜΠ. Αν ήταν και κλεισμένο των θυρών η συνεδρία, θα έλεγα ότι η επιλογή του υποψηφίου αιτιολογήθηκε ή κινήθηκε από το να υπάρχει μεγαλύτερη ε, αυτονομία από την εποχή, να ε, μην έχουμε καλές σχέσεις, αλλά ο καθένας να μπορεί να προασπίσει τη θέση του και τις απόψεις του. Και εμείς θέλουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα να προωθήσουμε. Για να μην είμαστε υποτελείς κανενός. Σε ό,τι αφορά τις μελίτες αντικτύπου, Εν συντομένα, φέρθηκα Πράγματι, αξίζει να πούμε ότι μέχρι τώρα, επειδή δεν ήταν ξεκάθαρο μέχρι τώρα, η μελέτη αντικτύπου μπορεί να φαίνονταν ανεπαρκής. Γι' αυτό και επέμεινα στο γεγονό ότι οι μελέτε αντικτύπου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα μακροοικονομικά στοιχεία και να πηγαίνουν πιο πέρα στην τοποθέτησή τους. Δεν είπα ότι η ΕΦΡΑΚ θα κάνει βέβαια πολιτική, δεν το πιστεύω αυτό, αλλά ένα σύμβουλο, μια συμβουλευτική επιτροπή, γιατί εγώ έχω διατελέσει σύμβουλο όταν είμαι δικηγόρο. Η ΕΦΡΑΚ θα πρέπει να λέει ποιο είναι ο κανόνα και τι πρέπει να γίνει, αλλά τελικά τουλάχιστον να γνωμοδοτεί. Μπορεί να, μάλλον δεν θα πρέπει να πει ποιο είναι ο κανόνα, θα πρέπει να δίνει μια συμβουλή, επειδή έχει μελετήσει σε βάθο ένα φάκελο, έχει ακούσει του μεν, του δε και αυτή είναι μια μέθοδος που θα ήθελα να προωθήσω. Με την ε, συνεργονόηση βέβαια και τη συνεργασία μου με τον Διευθυντή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Μπέρντ Λούκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω εκ μέρους ε, του κύριου Καμάλ, ο οποίος ε, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρόν. Χαιρόμαστε που ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλια που κάσαμε μέχρι τώρα. Εμείς ως ECR ε, θεωρούμε ότι ο διορισμός σας είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος, ε, ο οργανισμός τώρα αυτός υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι οι συστάσεις σας ε, έτυχαν ομόφωνης αποδοχής ε, και προσβλέπουμε σε περαιτέρω διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Είναι καθοριστική σημασία για μας η ΕΦΡΑΚ να προσφέρει τεχνική ανάλυση ψηλοεπιπέδου και ουσιαστική δέσμευση ε, έτσι ώστε ε, οι προδιαγραφές να προστατεύουν και να υπηρετούν το κοινό καλό. Να σας πω επίσης ότι χαιρετίζω αυτά που είπατε, ότι θέλετε να συνεχίσετε τη σχέση με το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να ε, διευκολυνθεί η συζήτηση που εξακολουθεί να λαμβάνει η χώρα ε, για τις ε, προδιαγραφές. Τώρα μπαίνουμε σε δύσκολη φάση της αξιολόγησης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κύριε Γκοζές ε, την άποψή σας για ένα θέμα ε, το οποίο τέθη σε μια πρόσφατη έκθεση για την αντίφαση σχετικά ε, με αυτά που λέει η ASB για τους λογαριασμούς και την περίπτωση της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε γιατί το θέμα τέτοι ήδη από τον Ζερόμ Haas από τη γαλλική πλευρά. Στην άποψη του ISB, ο στόχος των λογαριασμών ε, είναι να κρίνεται από ένα μοντέλο ε, το οποίο έχει και σχέση με τις κεφαλαγορές με στόχο να λαμβάνονται αποφάσεις για το πού θα ε, διανέμεται και πού θα δίδεται το κεφάλαιο. Με βάση τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για όλες τις απαιτήσει και τέτοιου είδους διατάξεις πρέπει να είναι γνωστές και να μην προσμετρώνται σε απώλειες. Μόνο τα κέρδη που βρίσκονται στους λογισμούς θα πρέπει να κατανέμονται ως μερίσματα. Αυτό αναφέρεται και στη σχετική οδηγία. Το ερώτημά μου είναι, εσείς αυτό το αναγνωρίζετε ως αντίφαση και εάν ναι, μήπως έχετε κατά νου κάποιο τρόπο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας, για την ερώτησή σας. Έλεγα πριν από λίγο ότι μπορεί να είναι υπερβολικά φιλόδοξη η ψηφιότητά μου, ίσως όμως θα ήταν ακόμη πιο φιλόδοξο να προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτό σας το περίπλοκο ερώτημα όπου δεν έχω την νομιμότητα, να επικρίνω δηλαδή οποιονδήποτε, οποιαδήποτε απόφαση άλλου οργανισμού. Αλλά βεβαίως ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, αυτή την ερώτηση αντικείμενο μιας, ενός πραγματικού προβληματισμού ώστε να μην ε, τα κάνουμε όλα αυτά στο πόδι ε, με τεχνικά στοιχεία για να σας προτείνω λοιπόν να ξαναβρεθούμε για να το συζητήσουμε με τους αρμόδιους, με ένα μικρό κύκλο αρμόδιων ανθρώπων, ώστε να δούμε ποιες, ε, ποια συμπεράσματα μπορούμε να αποκομίσουμε. Δεν ναι, σας απάντησα για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, κυρία Μπερέζ. Ε, φυσικά και με προβληματίζει. Είναι ένα, κάτι που με προβληματίζει από όταν ήμουν ευρωβουλευτής, αλλά θα ήθελα επίσης οι λογιστικοί κανόνες να μην τιμωρούν το είδος αυτό δραστηριότητας και μάλιστα όχι τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις λόγω μέτρων τελείως βραχυπρόθεσμων όπως η υπόθεση Βιολού, όπως και άλλες, ε, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Ευχαριστώ. Η Σιλβή Γουλάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να είμαι εδώ πίσω, γιατί έβαλα εδώ το, στην πρίζα τον υπολογιστή μου. Δεν είχα πρίζα πιο κοντά. Εδώ πίσω-πίσω. Γαλαρία. Ε, νομίζω πως ε, όντως θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την εξέταση πολύ σοβαρά αν και όλοι έχουμε εξαιρετικές αναμνήσεις από το πέρασμα σας από εδώ και για τις ε, ε, ικανότητές σας και τα προσόντα σας. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας όμως σε αυτή την θέση ε, βράχη πρόθεσμα και πιο μακροπρόθεσμα. Ίσως πιο μακροπρόθεσμα να μπορούσαμε να το συζητήσουμε ενδεχομένως, ε, αλλά θα έλεγα από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε σε αυτό το τομέα ε, πώς και όπως είπαμε και πρόσφατα σε μια έκθεση πρωτοβουλίας, ε, πώς ε, θα γίνει αυτός ο συσχετισμός, χωρίς να θέλω να σας παγιδεύσω, Α, είναι η προτεραιότητα, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του νεοδιοριστέντος Προέδρου. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, την έκθεση του κυρίου Στόλογιαν τη διάβασα με πολύ προσοχή. Διάβασα επίσης τις διάφορες τροπολογίες που διατύπωσαν ε, διάφοροι, ε, ε, ε, γιατί αυτά φωτίζουν με τον τρόπο το πώς το Κοινοβούλιο βλέπει τα πράγματα. Οι, δικέ μου, οι δικές μου προτεραιότητες, αν γίνω πρόεδρος, καταρχήν θα είναι να λειτουργήσει αυτή η ομάδα σε άμεση σχέση με το Γενικό Διευθυντή, γιατί οι περιστάσεις ε, οδηγούν στο ότι η ΕΦΡΑΓ θα έχει ένα νέο πρόεδρο, αφού δεν είχε, και έναν γενικό διευθυντή που είναι, εδώ, που είναι εκεί στη θέση του μετά από τη 11 Απριλίου. Δύο νέοι άνδρες. Καινούργιοι άνδρες, όχι νέοι. Αυτό ίσως να είναι ένα του, στο βαθμό που τελικά μπορεί να έχουμε νέες ιδέες χωρίς να είμαστε φυλακισμένοι οι όμοιροι των όσων έγιναν παλιότερα. Προτεραιότητα λοιπόν είναι να λειτουργήσει αυτή η ομάδα με αρμονικό τρόπο και το ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό. Είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλη αξία, μεγάλες ικανότητες και θα πρέπει να περάσουμε στις απαντήσεις και στις ε, ανταπόκριση προσδοκίας ε, που προκλήθηκαν μέσω της ε, απάντησης αυτής και της μεταρρύθμισης της ΕΦΡΑΓ. Και αυτό με την έννοια να έχουμε περισσότερη αποδοτικότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχω την αίσθηση σήμερα, και αυτό βέβαια είναι προσωπική μου αίσθηση, ότι ορισμένοι οργανισμοί κάπως έχουν μείνει πίσω ή δεν συνεργάζονται τόσο πολύ με τους υπολείπους όσο θα θέλαμε. Προβλέπω λοιπόν να έρθω σε επαφή πολύ σύντομα με τους τρεις προέδρους που ευτυχώς τους γνωρίζω γιατί ήταν ευρωβουλευτές ε, και ήμουν εγώ ευρωβουλευτή, συγγνώμη, όταν ορίστηκαν, όταν διορίστηκαν και θα έχω έτσι εύκολα, εύκολα πρόσβαση σε εκείνους και πάλι. Έπειτα έχουμε εκπροσώπους των εθνικών ε, ρυθμιστών. Και με εκείνους πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δουλέψουμε με τρόπο ώστε καλύτερα να αναπτύξουμε την δυνατότητα προπίσης σε σχέση με τις μικρομεσαίες που είναι μια ιδέα που θέλουμε να μπει παντού τη βλέπουμε και στην δική σας έκθεση του κυρίου Στόλογεν και ε, είναι μια δουλειά που πρέπει να την κάνουμε ώστε να παγιωθούν οι λογιστικοί κανόνες. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μου και για τα υπόλοιπα νομίζω ότι οι περιοδικές επαφές που προτείνω ε, να δουλέψουμε σε μια ομάδα που ενδιαφέρεται για αυτά τα ζητήματα, θα μπορέσουμε έτσι να τα ορίσουμε και να τα συζητήσουμε μαζί. Ε, νομίζω πως έτσι θα έχουμε καλά αποτελέσματα, αν δουλέψουμε όντως με συλλογικό τρόπο. Σας ευχαριστώ, Μακάρτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να μεταφέρω τη συγγνώμη του Φάμπιου Ντεμάς που δεν μπορεί να παραστεί. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει σχέση με τη σύνθεση των μελών στον ERSB. Να ρωτήσω κατά πόσον θεωρείτε ότι εκφράζονται και εκπροσωπούνται όλες οι διαφορετικές ομάδες, συνδικάτα, καταναλωτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργοδότες και όσον αφορά τους ε, οργανισμούς ε, που καθορίζουν τα πρότυπα τα λογισμικά, πιστεύετε ότι εκφράζονται, εκφράζεται το δημόσιο συμφέρον και αν όχι, ε, ποιο κρίνεται ότι τι κρίνουν ότι πρέπει να βελτιωθεί. Και το δεύτερο σκέλος ερώτησή μου είναι προσωπικό. Πολλοί από εμά πιστεύουμε ότι ένα τμήμα της κρίσης της οικονομικής ε, οφείλεται στη συνένεση που ήταν απαραίτητη για την προστασία των θεσμών σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους πολίτες. Ξέρω ότι έχετε υπηρετήσει εδώ πολύ καιρό, ότι έχετε εμπλακεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο ευρωπαϊκό πολιτικό οικοδόμημα. Ακούω ότι έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό. Εσείς μπορείτε να με καθησυχάσετε ότι δεν είσαστε κι εσείς σε ένα σύστημα αυτών των ε, ανακυκλούμενων θυρών, δηλαδή των ανθρώπων που μεταπηδούν από τη μία θέση στην άλλη. Και ε, θα ήθελα με πολύ μεγάλη μου χαρά να σας ακούσω να με καθησυχάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Για την οργάνωση του ΕΦΡΕΚ. Θα κατανοήσετε ότι όταν είμαστε υποψήφοι σε έναν οργανισμό που υπάρχει και που πρόσφατα μεταρρυθμίστηκε και για τον οποίο δεν μπορέσαμε ακόμα να αξιολογήσουμε τις συνέπειες αυτής της μεταρρύθμισης, δεν θέλω να λάβω θέση για την σκοπιμότητα της σημερινής οργάνωση της ΕΦΡΑΓ. Θα ήταν ε, μάλλον ε, ε, Άτοπο και δεν αντιστοιχεί στις στην υπευθυνότητα. Την κατάλληλη στιγμή ε, οι αρμόδιες αρχές ε, θα μπορέσουν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς και της μεταρρύθμισης. Αλλά δεν είναι τώρα δική μου δουλειά να κάνω παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ε, λειτουργήσε το κοινοβούλιο. Βρίσκω πως το ΙΦΡΑΓ και η ιδέα ενός οργανισμού που αντιπροσωπεύει διαφορετικά και διάφορα συμφέροντα είναι καλή ιδέα, Ορισμένοι θα ήθελαν να είναι δημόσιος αυτός ο οργανισμός. Δεν ε, ε, έγινε δεκτή αυτή η πρόταση. Εγώ λοιπόν εντάσσομαι στο νομικό πλαίσιο και αν κάποιος, κάποιοι θεωρήσουν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, εγώ δεν θα φέρω αντίρρηση, θα τις εξετάσω και θα ενεργήσουμε αναλόγως. Τώρα, 2000 9 μέχρι 2014. Εργάστηκα πολύ για οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα και ε, συμφωνώ με την εργασία που έγινε από την πλειοψηφία σε αυτή τη φάση. Ήταν μια πλειοψηφία ευρύτατη που είχε συνείδηση για το ότι η κρίση ήταν έντονη και ότι έπρεπε να υπάρξουν ε, διορθώσεις. Ε, ίσως οι διορθώσεις αυτές δεν ήταν τέλειες, αλλά σίγουρα ήταν λιγότερο κακές από το να μην γίνει τίποτα και υπήρξαν και κάποιες οριοθετήσεις και αυτή η εργασία είναι γενικά θετική. Κατά τα λοιπά σας διαβεβαιώ ότι δεν ανήκω σε κανένα μυστική, καμία μυστική οργάνωση και αν θέλετε να πάτε και πιο μακριά όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, από τότε που δεν είμαι πια βουλευτή, ευρωβουλευτή, δηλαδή εδώ και δύο χρόνια, δεν έχω ασχίσει καμιά αμοιβόμενη λειτουργία και καμία συμβουλευτική λειτουργία και έχω αρνηθεί όλες τις προτάσεις που μου επιβλήθησαν για να κάνω λόμπινγκ. Είμαι απλά ταμείας. Θα έλεγα κανείς ότι έχει λεφτά εκεί, αλλά δυστυχώ δεν έχει. Είμαι ταμείας του Ιδρύματος Σούμαν, που είναι ένα ίδρυμα κοινοφελέ που προσπαθεί να προωθήσει τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Τώρα, άμα θέλετε αυτό να πείτε ότι είναι δέσμευση, ναι, η Ευρώπη είναι δέσμευσή μου. είναι γκολτ. Σας ε, καλωσορίζουμε θερμά. Ζαμπόλ, ε, επειδή μιλάς ε, πάρα πολύ καλά γερμανικά, θα μιλήσω και εγώ λιγάκι γερμανικά, γιατί και οι συνάδελφοί μου αμφισβητούν πια αν μπορώ να μιλάω γερμανικά. <laughs> αγαπητέ Βέρνα, εσύ που έρθες και από την Ανία Παλατινάτο, θα πρέπει να προσέχεις λιγάκι με τη διάλεκτο που μιλάς. Λοιπόν, τώρα αυτά για γερμανικά, μιλάω αγγλικά. Νομίζω ότι είναι ένδειξη σοφίας από πλευράς Επιτροπής, το ότι σε προτείνανε ως υποψήφιο και νομίζω και είναι μια ένδειξη της ε, αυξανόμενης επιρροής ε, που ασκεί το Κοινοβούλιο στον ε, λογιστικό τομέα. Είναι η δεύτερη φορά που ένας πρώην συνάδελφος ορίζεται και προτείνεται για αυτό τον τομέα. Εγώ επιθυμώ η ΕΦΡΑΚ να εξετάζει περισσότερο τις μακροοικονομικές δυνατότητες και επίσης μου άρεσε αυτά που είπατε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τη δημοκρατία, για τη λογοδοσία της ΕΦΡΑΚ στο Κοινοβούλιο και τέλος ε, και τις θετικέ αναφορές στην έκθεση Στόλογιαν. Νομίζω ότι ε, υπήρξε μακρά συνεργασία εδώ, ε, ξέρουμε πώς μπορούμε να σε δούμε. Μία ερώτηση είναι η έκθεση Ντελαρουζιέρ που ήταν το σημείο κίνησης για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη. Στην έκθεση Ντελαρουζιέρ, όπως και στην έκθεση Στόλογιαν, υπάρχουν πολλές αναφορές ε, στους ε, κανόνες ε, λογιστικής και η αμοιβαιότητα που μπήκε σε αυτούς τους κανόνες προκάλεσε την κρίση. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα ε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συνέπειες από όλα αυτά. Εσείς προτίθεστε να επανεξετάσετε αυτό, αυτή την κληρονομιά, την παρακαταθήκη του Ντελαροζιέρ. Επίσης λέτε ότι πρέπει να υπάρχει πιο ισχυρή Ευρώπη στα λογιστικά πρότυπα, με δημοκρατία, με αξίες. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αυτά πρέπει να ισχύουν και στους διεθνείς οργανισμούς, ότι θα ισχύουν οι δημοκρατικές αρχές. Και τέλος, ε, θέλετε να μας δώσετε έναν κατάλογο όλων των ε, εκπροσώπων λόμπις που σας πρόσφεραν δουλειά. Äh, <laughs> Μπορώ να σας δώσω τον κατάλογο, δεν και πολύ. Δεν έγινε και ουρά όπως γίνεται στα Πενιζινάδικα σήμερα, αυτές τις μέρες τέλος πάντων στη Γαλλία, μπροστά στο γραφείο μου, αλλά για το πρώτο σου ερώτημα, ό,τι έχει να κάνει με τη δημοκρατία. Ε, είδες, θα μιλήσω και γερμανικά σε λίγο. Είμαι ανοιχτός να γίνει κάποια συζήτηση ε, και να τεθεί επιτάπητο στο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τα στοιχεία τα προκυκλικά. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία πιστεύω και εγώ ότι έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, είχαν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην κρίση. Και όταν ε, μιλούσα για ένα ενεργητικό ρόλο της ΕΦΡΑΚ, των προτέρων να δραστηριοποιούμαστε, μιλούσα ακριβώς για αυτές τις συνομιλίες και τις συνεννόησεις μεταξύ Κοινοβουλίου και ΕΦΡΑΚ, ώστε να ξαναθέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα επιτάπητος και να δούμε ποιες τεχνικές δυνατότητες υπάρχουν. Γιατί είναι ενδιαφέρον για την έφρακα που είναι ένας ε, τεχνισμός ε, οργανισμός με μεγάλη τεχνική εμπειρία, να μπορούμε να δώσουμε κάποια στοιχεία απάντησης και να έρθουμε τελικά με λύσεις που θα μπορούσαν να συζητηθούν από τους διάφορους φορείς, αλλά να έρθουμε με κάποιες ε, ιδέες αρχικές για συγκεκριμένες λύσεις. Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι αν με εμπιστευτείτε θα προσπαθήσω να ασκήσω την Προεδρία με κοινωνού. Αυτό λένε ότι είναι γαλλικό χαρακτηριστικό, δεν το ξέρω αυτό, και με ρεαλισμό πραγματισμό που λένε ότι είναι βρετανικό χαρακτηριστικό. Αλλά σίγουρα θα ενεργήσω με βάση το δημόσιο συμφέρον. Αυτό είναι ο στόχο μου. Αλλά ο στόχο αυτό δεν θα επιτευχθεί παρά ε, χάρη και στην ποιότητα τη ομάδα τη ΕΦΡΑ και είναι κάτι που δεν αμφισβητώ και χάρη και στη σχέση εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ τη ομάδα τη ΕΦΡΑ και του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Το FTD μήπως θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Δεν έχω κάποιον ομιλητή από εσά. Στην ομάδα το ENF μπορούμε δηλαδή να ολοκληρώσουμε την ακροασία μας σε αυτό το σημείο. Εξαιρετικά. Σας συγχαίρουμε. Και τώρα χρειάζεται πάρα πολύ σύντομα πιστεύω εμείς να κάνουμε την εικασιολόγησή μας ε, και να ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκοζές. Και κλεισμένο των θυρών τώρα, αλλά για πολύ σύντομα ε, για να κρίνουμε την υποψηφιότητα όσοι δεν επιτρέπεται να μείνουν παρακαλώ να φύγουν από την αίθουσα για να έχουμε την συνεδρίασή μας και κλεισμένο των θυρών παρακαλώ να αποχωρήσετε όσοι δεν έχετε εργασία και εκείνο ο ίδιο μπορεί να έρθει. Α, όχι. Πρώτα να ψηφίσουμε και μετά να τον συγχαρούμε. Πρέπει να γίνει ένα, μια δοκιμή. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε ναι και, στο, στη δοκιμή. Δοκιμή κάνουμε τώρα. Δύο ακόμη πρέπει να ψηφίσουν. Okay, the vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Τέλεια. Τώρα, επίσημα τώρα ψηφοφορία άρχεται. Η ψηφοφορία για το διορισμό του Προέδρου του ΕΦΡΑΓ. Τι είναι μυστικό. Ναι, Μυστική ψηφοφορία. Secret ballot. Okay. So now, so... Ωραία λοιπόν. Δεν ήταν μυστική ψηφοφορία έτσι κι Λοιπόν, ο κανόνας είναι... Τώρα είναι όμως μυστική. Γιατί ο κανονισμός λέει να είναι μυστική. The is Τέλος της ψηφοφορίας. Μάλιστα. 36 υπέρ. 5 κατά. 2 αποχές. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον κύριο Γκουζέση. Και τώρα προχωράμε στη ψήφο μη αντίρρησης. Όπως ξέρετε, Υπάρχει μια πρόταση να βάλουμε μία αντίρρηση στην πρόταση 596 για την κατάχρηση της αγοράς από πλευράς της Κομισιόν. Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε unblock το αρχικό κείμενο. Ψηφίζουμε. Τώρα αυτό δεν είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται. Πέρας. 37 υπέρ. 6 εποχές εγκρίνεται. Thank you. Next meetings. Uh, Ευχαριστώ. Επόμενη συνεδρίαση 30 Ιουνίου. Πέρα συνεδρίαση. 13 of June. 13 εννοούσε ο πρόεδρος. 13 όχι 30, ναι. Σε 13 μέρες, ναι. We will be happy on 13 to see again each other.